Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι, οπότε το αίτημα αυτό εγκρίνεται. Και τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε την πρώτη μας συζήτηση για την περίπτωση παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Η πρώτη συζήτηση για απόψε αφορά το Ιράν και τις προς, τα πρόσφατα περιστατικά παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δίνω το λόγο στον κύριο Μπέλντερ για 2,5 λεπτά. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την ώρα, η ζωή του Ιρανού ε, παπά Γιούσεφ Αραχάνη είναι, εξαρτάται από την κρίση του Αγιατολάχ Χαμενή, που είναι ο ανώτατος δικαστής και ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Θανατική ποινή του έχει αποδοθεί λόγω αποστασίας. Γιατί θέλησε να αλλαξοπιστήσει. Και αυτή είναι μια καταδίκη που περιλαμβάνεται στο Ιρανικό Σύνταγμα, στην ποινική νομοθεσία, αλλά είναι αντίθετη προς τις διεθνείς συνθήκες, διεθνείς συνθήκες ε, τις οποίες έχει συνυπογράψει το Ιράν. Για πολλούς ε, θα μπορούσε, ο Χαμένη θα μπορούσε να απελευθερώσει τον Αντραχάνη, ε, είναι μια πιθανότητα αυτή, ωστόσο έχουν έχει υποθεί πολλές φορές, αλλά ποτέ δεν έχει γίνει. Γι' αυτό και ο κόσμος φοβάται ότι θα υπάρξει δραματική τροπή στην υπόθεση κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων δικοπών. Παρακαλώ, συνάδελφοι, λοιπόν, μην αφήσετε να πάει ο Ναντερκάνη στην Αγχώνη. Ζητήστε την απελευθέρωσή του από τις Ιρανικές αρχές. Ε, ένας Ιρανός ε, δημοσιογράφος μου τηλεφώνησε χθε το βράδυ πολύ αργά και ακόμα ακούω τη φωνή της τα αυτιά μου. Γιατί η Ευρώπη σιωπή κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί είναι τόσο παθητική δεδομένου ότι η ζωή του να ε, είναι ε, κρέμεται από μια πολύ λεπτή κλωστή. Μιλάμε για ένα πολύ επίκαιρο θέμα και θα θέλαμε να δώσουμε μια αξιοπρεπή ανθρώπινη απάντηση. Και φυσικά αυτό ισχύει για κάθε παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων που θα συζητήσουμε σήμερα και σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κύριε Μπέλντερ. Η κυρία Βεργιά είναι η επόμενη. Merci, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εξετάζουμε σήμερα ένα ψήφισμα για το η Ιράν για έκτη φορά από την αρχή της θητείας μας. Τρίτη φορά μέσα στο 2011. Συμφωνώ με το περιεχόμενο του ψηφίσματος. Μια φορά ακόμα όμως θα ήθελα να επιμείνω ε, στο όραμά μας. Παντού στο όλο τον κόσμο, γυναίκες, άντρες και παιδιά ε, συλλαμβάνονται, δικάζονται, ε, και πολλές φορές θανατώνονται ε, και εμεί σιωπούμε. Να σας πω το εξής παράδειγμα. Σήμερα το πρωί ένα νέο Τινήσιο, 27 ετών, εκτελέστηκε στο Ιράκ. Μέχρι τελευταία στιγμή φώναζε την αθωότητά του και είπε ότι η ομολογία του το με βασανιστήρια. Ο πρόεδρος του Ιράκ ενέκρινε αυτή την θανατική ποινή. Ε, αυτή η χώρα, ε, το κοινοβούλιο, στο κοινοβούλιο, ε, το κοινοβούλιο αυτής της χώρας δεν έχει ψηφίσει τίποτα από τον Ιούλιο και μετά. Η κυρία Κρέτου, παρακαλώ. Μιλάμε ξανά για το Ιράν και τα όσα γράφει το ψήφισμα επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες μας. Το καθεστώς με τη βία προσπαθεί να καταπνίξει τις αντιδράσεις του πληθυσμού. Ε, οι Ιρανικές αρχές ε, καταχρώνται της εξουσίας τους ε, και επιτίθενται εναντίον μειονοτήτων, γυναικών, παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλοι οι υπεύθυνοι ε, μάλλον όλοι οι αντιδρόντες ε, τιμωρούνται. Η διεθνής κοινότητα έχει εκφράσει τις ανησυχίες της ε, για τα, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν επανειλημμένως. Το Ιράν απάντησε με περισσότερη βία και περισσότερη καταπίεση, περιορίζοντας ακόμα περισσότερο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι Ιρανικές αρχές θα πρέπει να δείξουν λογική και να απονείμουν δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπίλαν, η δίωξη της αντιπολίτευσης και η, η καταπίεση ε, με βάση τα θρησκευτικό ε, πιστεύω αξίζουν την καταδίκη από πλευράς μας. Έχουμε πολλές περιστατικά όπως η Ρεζίλτα Φάρμαρ που ε, είναι καταδικασμένη και έχει μαστιγωθεί επειδή έφτιαξε αυτό το, την ταινία. Ε, οι χώρες ωστόσο προβαίνουν σε οικονομικές σχέσεις με το Ιράν ανεξάρτητα από την αντιμετώπιση των αντιρρησιών συνείδησης συμπεριλαμβανομένου του Νανταρκάνη. Εγώ θέλω να κάνω έκκληση για να ασκήσουμε πιέσεις μέσω συντονισμένων κυρώσεων. Να αναγκαστούν οι αρχές της Τεχεράνης να συνεργαστούν με τον ΟΗΕ και να υποστούν έλεγχο σε ολόκληρη τη χώρα. Ο κύριος Πρέντα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα λεπτό είναι πολύ λίγο για να αναφέρει κανείς μια ολόκληρη σειρά παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Πρόκειται για συλλήψεις, για αυθαίρετες κρατήσεις, για συνοπτικές ε, δικαστικές διαδικασίες, για βασανιστήρια, για παραβίαση των ανθρωπίνων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και για την θανατική ποινή. Ξέρουμε ότι η παγκόσμια τάση είναι προς την κατάργηση της θανατικής ποινής. Πολλά ψηφίσματα του ΟΗΕ έχουν ζητήσει μορατόριο διεθνές, ωστόσο το Ιράν παραμένει το κράτος το οποίο έχει το, τις περισσότερες θανατικές ποινές σε σχέση με τον αριθμό του πληθυσμού και πολύ συχνά οι εκτελέσεις γίνονται με απόλυτη μυστικότητα. Η έκθεση λέει 300 μυστικές εκτελέσεις πέρσι και συχνά είναι ανήλικη τα θύματα. Ο συνάδελφος ζήτησε άμεση απελευθέρωση του πάστορα Ιουσέφ Νανταρκάνη, ο οποίος κατηγορήθηκε για αποστασία επειδή προσιλητήστηκε στο χριστιανισμό πολύ νέος. Πιστεύω πως ε, οι σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ιράν θα πρέπει να αναθεωρηθούν ακριβώς για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Κύριε Σάκε, από πού να ξεκινήσει κανείς. Το πυρηνικό θέμα βρίσκεται στην κορυφή της ε, ε, ατζέντα μας, τη ημερησίας διάταξης, αλλά μην ξεχνάμε ε, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα ενώπιον των εκλογών της Άνοιξης που έρχεται. Αυτή τη στιγμή καταπιέζουν οι πολίτε, εκπαιδεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα δικαιώματα των γυναικών, καταπιέζεται ε, ο τύπο, τα μέσα ενημέρωση, ψηλότατο δείκτη θανατικών ποινών, πιο ψηλό και ακόμα και από τη Κίνα, ε, συμπεραμένων και παιδιών. Ε, ε, και βέβαια βία και βασανιστήρια. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε του γενναίου Ιρανού. Βέβαια το μέλλον της χώρας βρίσκεται στα χέρια του λαού της και είμαι σίγουρος θα τα καταφέρει. Αλλά ακόμα και με τις κυρώσεις του ΟΗΕ ε, οι ευρωπαϊκές εταιρείες εξακολουθούν να παρέχουν βοήθεια ε, μέσω της ε, τεχνολογίας που διαθέτουν και της τεχνονοσίας τους για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό πολιτών του Ιράν. Θα πρέπει να σταματήσουμε να βοηθάμε με τέτοιου είδους τεχνολογία το Ιρανικό καθεστώς. Οι κανονισμοί διπλής, προϊόντων διπλής χρήσης δεν αρκούν. Χρειάζεται να υιοθετήσουμε ένα μηχανισμό αδειοδότησης πριν από τις εξαγωγές και δεύτερον ε, έναν, ε, ένα σχεδιασμό έτσι ώστε ε, οι ευρωπαϊκές εξαγωγές να μην πλήττουν τον Ιρανικό λαό. Ευχαριστώ κύριε Λόχ Ευχαριστώ πρόεδρε. Πραγματικά οι τίτλοι των διεθνών εφημερίδων αυτές τις μέρες συγκεντρώνουν την προσοχή τους στο πυρηνικό πρόβλημα. <clears throat> Είναι καλό που εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, έχουμε κατά νου στο επίκεντρο να θέσουμε το θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που όσο πάει και επιδεινώνεται. Το ψήφισμά μας έχει σαν στόχο την απαρίθμηση των πολυαρίθμων και σοβαρών καταπατήσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους οποίους εκτίθονται οι πολίτες του Ιράν. Είναι φρικτή, φρικτός ε, και ο κατάλογος αυτός. Παραδείγματο χάρη να αναφέρομαι εδώ στο ταπεινωτικό μαστίγωμα φοιτητών και ζητάμε ο ποινικό κώδικας του Ιράν να τροποποιηθεί για να αποφεύγονται αυτού του είδους οι τιμωρίες σε μια ενδιάμεση έκθεση η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφέρθηκε σε επιδεινούμενη κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα συστηματικό πρότυπο βίας και καλούμε την ε, Ιρανική κυβέρνηση να λάβει σοβαρά υπόψη αυτή την έκθεση και να επιτρέψει σε έκτοξου απεσταλμένου την επίσκεψη επιτόπου. Το ψήφισμά μα έχει όμω σαν στόχο και επιχειρήσει που έχουν έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και που πουλούν ε, τεχνογνωσία και εξοπλισμού στο Ιράν. Ε, τεχνολογία με την οποία ε, το Ιράν πολλές φορές διώκει τους πολίτες του και ε, τους, ε, το χρησιμοποιεί και επίσης για την επιβολή βασανισμών. Θα πρέπει σύμφωνα με τις Ισλαμικές αρχές να υπάρχει ένα δίκτυο χαλάλ λέγεται, αλλά αν το εξετάσει κανένας προσεκτικά βλέπει ότι αυτό είναι ένα μέσο για να ελέγχεται ο πληθυσμός, επιτρέπει όμως ε, εξαιρέσεις. Και επικρίνω ότι από την Ευρώπη εξάγονται τεχνολογίες και φίλτρα στο Ιράν. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό γιατί αλλιώς έχουν συν ε, ευθύνη για την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και παρακαλώ όλους τους συναδέλφους να υπερψηφίσουν τις σχετικές μας τροπολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ εγώ. Θα ακούσουμε τώρα τις πολιτικές ομάδες, αρχίζοντας με το ΕΛΚ, την κυρία Μακοβέη το Ιράν είναι μία από εκείνες χώρες στις οποίες κατά τον 21ο αιώνα οι πολίτες εξακολουθούν να διώκονται από τη δικαιοσύνη και είναι αναγκασμένοι να κάνουν την επιλογή μεταξύ του θρησκευτικού τους πιστεύω και της ζωής τους. Αυτό βλέπουμε ακούγοντας τον ε, η ιερέα Κουγανταζή, ο οποίος καταδικάστηκε σε θάνατο διαποχωνισμού. Ο μεγάλος αριθμός των εκτελέσεων και δημοσίων εκτελέσεων και με λιθοβολισμό, οι βασανισμοί, η βιότητα των τιμωριών, το τυχαίο των ε, αποφάσεων ο σοβαρός περιορισμός της ελευθερίας έκφρασης και συνέχεστε είναι ανησυχητικά μηνύματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Λυπούμε για την απόφαση της Δευτέρας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων που ανέβαλε την ε, ε, επιδείνωση των ε, κυρώσεων κατά του Ιράν. Χρειαζόμαστε πιο ε, ευρεία συνένεση την επιτρέπει να πραγματοποιούμαστε το σεβασμό θρήμα δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. εξ των Αυτό το ψήφισμα αναφέρει λεπτομέρειες για τις βάρβαρες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα βασανιστήρια και τις εκτελέσεις στο Ιράν. Αυτά λαμβάνουν χώρα συστηματικά εναντίον των πολιτών του Ιράν. Ε, με εκπλήσει ε, η μάλλον θαυμάζω την πολιτιστική κληρονομιά του Ιράν ε, και ε, προφανώς ε, η συμπεριφορά αυτή του καθεστώτος δείχνει το φόβο του. Άλλωστε το καθεστώς αρνείται να συνεργαστεί με τον εισηγητή του ΟΗΕ που έχει οριστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τη μεριά της πρέπει να κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει αυτούς που θαραλέα αγωνίζονται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Και είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η παρουσία ευρωπαϊκών εταιριών που προμηθεύουν ε, το καθεστώς του Ιράν τεχνολογία που τους επιτρέπει να εντείνουν τη λογοκρισία. Αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναδειχθούν ποιε είναι και να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάχη. Κύριε Πρόεδρε. Να είμαστε άλλη μια φορά εδώ, συζητώντα ε, την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τι παραβιάσει αυτών στο Ιράν. Είναι μια, ε, δρόμο. Ε, ε, ένας ατέλειωτος δρόμος Διαρκώ έχουμε στα κατεπήγοντα το Ιράν και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κόσμος του Ιράν αξίζει ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία και τη δημοκρατία. Ωστόσο, οι ακτιβιστέ ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικών δικαιωμάτων κρατώνται. Οι δικαστικέ διαδικασίες πολύ απέχουν από τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Τα δικαιώματα των γυναικών δεν γίνονται σεβαστά και η αρχή της ελευθερίας έκφρασης παραβιάζεται καθημερινά. Εγώ πραγματικά ε, Είμαι εξοργισμένη γιατί οι 42 δικηγόροι έχουν ε, διωχθεί και έχουν ε, και αυτή τη στιγμή κρατώνται γιατί προσπάθησαν να στηρίξουν πολιτικούς ακτιβιστές. Κύριε Πρόεδρε, η Αραβική Άνοιξη έδειξε ότι ο αγώνας των, ανθρώπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ελευθερία είναι ε, πάντα πολύ έντονος. Ε, εύχομαι ότι ο Ιρανικός λαός σύντομα θα υψώσει τη φωνή του και θα διεκδικήσει τα δικαιώματα που το αξίζουν. μεταξύ η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ε, διατηρήσει το θέμα αυτό ψηλά στην ημερήσια της διάταξη. Σας ευχαριστώ κυρία Γιατανμάκη και τώρα ο κύριος Βαντάλεν. Στο Ιράν κανείς πια δεν νιώθει ασφάλεια. Ε, γίνονται εκτελέσεις, γίνονται λιθοβολισμοί ε, και ε, από όλους τους Ιρανούς οι πιο ευάλωτοι είναι οι χριστιανοί. Φέτος ο Αχμαντίνε Τζάντ ξεκίνησε με ολόκληρη εκστρατεία εναντίον των χριστιανών με σλόγγαν «Ας δώσουμε τέλος στην ε, εξάπλωση του χριστιανισμού στο Ιράν. Και αυτό δεν αποτελεί μια απλή απειλή. Ο Ιουσέφ Νανταρκάνη βρίσκεται φυλακισμένος εδώ και δύο χρόνια και έχει καταδικαστεί σε θάνατο επειδή απαρνήθηκε το Ισλάμ και αποστάτησε, ε, προσιλητήθηκε στο χριστιανισμό. Ζητώ από την κυρία Δαμανάκη να πάρει αυστηρά μέτρα εναντίον του Ιράν ε, και η Ρωσία και η Κίνα θα πρέπει να μας υποστηρίξουν. Δεν θα πρέπει να περιοριστούμε μόνο στα λόγια, πρέπει να προχωρήσουμε σε πράξεις. στις, uh, τις, ε, τη μεγάλη καταπίεση που δέχονται, τις εκτελέσεις βασανισμού, τις φυλακίσεις, ο γενναίος λαός του Ιράν εξακολουθεί να κινητοποιείται μαζικά εναντίον του καθεστώτος όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Τελευταία έχουμε μια αύξηση του εργατικού κινήματος, δημιουργούνται ανεξάρτητα εργατικά συνδικάτα, ε, μαζικές απεργίες ε, στο, στην, ε, στον τομέα του ζαχαροκάλαμου, στο, στα πετρέλαια, στους, δα, στους δασκάλους, όλες αυτές οι κινητοποιήσεις ε, αντιμετωπίστηκαν με βία ε, και με φυλακής πολλών εργαζομένων. Η δικτατορία του Ιράν λοιπόν προβαίνει σε πολλές παραβιάσεις ανθρώπινων δικαιωμάτων ε, αλλά ε, δεν θα πρέπει αυτό να το χρησιμοποιήσουν ως αφορμή οι Ευρωπαίοι ηγέτες για να ε, επιβάλλουν κυρώσεις που θα βλάψουν το λαό ή να προβούν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αντιθέτως θα πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειές μας να καταδεικνύουμε κάθε φορά και να φέρνουμε στην επικαιρότητα τις παραβιάσεις αυτές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εργασιακών κινημάτων. Pan poslanec Πάσκα, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Το θέμα του Ιρανικού καθεστώτος έχει συζητηθεί επανειλημμένως, όμως οι εξελίξεις στη χώρα δείχνουν ότι η συμπεριφορά του φανατικού Ιράν γίνεται όλο ένα και πιο βίαιη. Η στάση απέναντι στις γυναίκες, τους ακτιβιστές, τους δικηγόρους, ακόμα και στα μέλη της οικογένειάς τους γίνεται διαρκώς πιο άγρια. Απλώς καταδιώκουν οποιονδήποτε εκφράσει οποιαδήποτε γνώμη κατά της δικής τους εξουσίας. Το θέμα του Ιράν νομίζω θα πρέπει να ακολουθήσει δύο δρόμους. Καταρχήν να καλέσουμε τις επίσημες Ιρανικές αρχές να σεβαστούν την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη εξωπρέπεια και την ε, ελευθερία λόγου και θρησκείας. Και το δεύτερο είναι να καταγράψουμε οποιαδήποτε περίπτωση εγκληματικής συμπεριφοράς ε, των Ιρανικών αρχών και να τα προσφέρουμε όλα αυτά στο Διεθνές Δικαστήριο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Σκέλη. Όταν μιλάμε για το Ιράν, απογοητεύεται κανείς απελπίζεται. Τα ανθρώπινα δικαιώματα και το Ιράν δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους και υπάρχουν εκατοντάδες ε, παραδείγματα. Η υπόθεση Ναντερκάν είναι η συγκεκριμένη που τονίζουμε σήμερα, αλλά μπορεί να εκτελεστεί ανά πάσα στιγμή για την κατηγορία αποστασίας από τη θρησκεία. Η πολιτική του Ιράν είναι ένα κράτος, μια θρησκεία. οποιοδήποτε δεν ασπάζεται το Ισλάμ κινδυνεύει να εκτελεστεί, να συλληφθεί οτιδήποτε ή να δυσκολευτεί. Άνδρας ή γυναίκα δεν έχει σημασία. Το Ιράν μόνο μπορεί να συναγωνιστεί την Κίνα. Είναι μπροστά από την Κίνα, 100 εκτελέσει το χρόνο. Παρά το γεγονός ότι το Ιράν έχει συνυπογράψει διεθνείς συμβάσεις και συμφωνίες που εγγυώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, νομίζω πως πρέπει πλέον να ενεργήσουμε πιο αυστηρά, πιο σταθερά ως ε, θεσμικό όργανο της Ένωσης και να στηρίξουμε τον λαό του Ιράν. Σας ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Ρέπο. Σας ευχαριστώ πρόεδρο. Ε, απαρίθμηση των παρεμβάσεων του Ιράν είναι πάρα πολύ μακρά. Τους τελευταίους μήνες Είδαμε ε, καλλιτέχνες, ε, ε, δικηγόροι και περιβαλλοντολόγοι να διώκονται στο Ιράν. Και επίσης γυναίκες βλέπουμε να διώκονται μια Μειονότητες εθνοτικές επίσης ξέρουμε ότι έχουν ε, εκτελεστεί και γυναίκες και έφηβοι και μένουν στις φυλακές κάτω από απάνθρωπες ε, ε, συνθήκες και μάλιστα και με βασανισμούς. Το Ιράν δεν τηρεί καθόλου τους διεθνείς του υποχρεώσεις όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό θα πρέπει να ε, παρουσιαστεί ξεκάθαρα, γιατί θα πρέπει το Ιράν να σέβεται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτή είναι η μόση καλή βάση για ισορροπία στην κοινωνία του Ιράν. Το Ιράν παίζει ένα κακό παιχνίδι γιατί δεν μπορούν να ανεχθούν όλα τα πράγματα αυτά. Τι. Κύριος Πορεύα, επανειλημμένος έχουμε κάνει έκκληση στις Ιρανικές αρχές ε, να δώσουν τέλος ε, στην καταπίεση κοινωνίας τους. Και ε, θα πρέπει να σταματήσει η καταπίεση ε, ο όλων όσων ε, δραστηριοποιούνται για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Τα, ε, τα αποτελέσματά μας όμως ήταν ελάχιστα μέχρι τώρα. Θα πρέπει να πιέσουμε το Ιρανικό καθεστώς, να συνεχίσουμε να το πιέζουμε και ασφαλώς ε, θα πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν ήδη κάποιοι ε, περιορισμοί εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκ μέρου ε, στελεχών του καθεστώτο και έχουν μπλοκαριστεί και πολλοί τραπεζικοί λογαριασμοί, αλλά θα πρέπει να ε, πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα έτσι ώστε οι Ιρανοί να μην μπορούν να προμηθευθούν τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να παρακολουθούν του πολίτε του. Σήμερα το Ιρανικό καθεστώς χρησιμοποιεί την βία ως ένα εργαλείο εξουσίας. Χρησιμοποιεί τη βία για να τιμωρήσει όσους είναι αντίθετοι προς το καθεστώς. Διαρκώς παραβιάζονται βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και πολιτικά δικαιώματα. Είναι απαράδεκτο, δεν υπάρχει ε, τίποτα που να μπορούμε να δεχτούμε. Και όλα αυτά συμβαίνουν στο Ιράν, ενώ συμβαίνουν ε, ε, ρηξικέλευτες αλλαγές στον υπόλοιπο αραβικό κόσμο. Νομίζω ότι αν επιμείνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ε, είναι κάτι το οποίο θα στηρίζει οποιαδήποτε λογική κοινωνία, άσχετα από τη θρησκεία της ή το, ε, ε, ιστορία της. Δεν μπορούμε να ανεχόμαστε αυτή την καταστολή, αυτή την κατοπίεση όσων αγωνίζονται για τα βασικά τους δικαιώματα. Εγώ στηρίζω αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κούτας. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο στρατόπεδο Ασράφ που βρίσκεται στο Ιράκ και που μένουν 3.400 αντικαθεστατικοί σε πολύ δύσκολες συνθήκες θα πρέπει να προστατευθούν ε, σύμφωνα με τον ΟΗΕ από τις διώξεις. Ε, όλα αυτά, ο Ιρακινός Πρωθυπουργό ανακοίνωσε ότι θέλει να κλείσει αυτό το στρατόπεδο, πράγμα που θα δημιουργήσει, θα προκαλέσει μια πολύ σοβαρή ανθρωπιστική κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό, ε, ο ορισμός, ο διορισμός ενός ε, ύπατο εκπροσώπου για το στρατόπεδο Αστράφ είναι κάτι πολύ το θετικό. Θα πρέπει αυτός να καταφέρει το κλείσιμο αυτού του στρατοπέδου να αναβληθεί για αργότερα. Η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες επίσης έχει το καθήκον να ε, χειριστεί όσο γίνεται καλύτερα την κατάσταση αυτών των ανθρώπων και να τους οικηθεί την ασφάλειά τους. Το μόνο, η μόνη λύση που μπορούμε να βρούμε σε αυτό το πρόβλημα θα πρέπει να είναι ειρηνική. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Έχω πιο, ε, πιο πολλά αιτήματα. Θα κάνω ό,τι μπορώ. Πρώτα απ' όλα η κυρία Γιορδάν. Πρόεδρε, χθε ακούσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο διάφορα για το συμβαίνοντα στα, στις φυλακές του Ιράν, στους δρόμους, στα σπίτια, στα πανεπιστήμια. Μια πολιτική έντονα κατά των γυναικών βλέπουμε να υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Θα ήθελα λοιπόν να επιστήσω την προσοχή σας στην ε, κατάσταση των προσφύγων στο στρατόπεδο Άσραφ που πρόκειται να κλείσει τέλη του έτους. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για τους ανθρώπους αυτούς. Θα πρέπει να κάνουμε κάτι για να τους φροντίσουμε. Η απόφαση αυτή της ε, κυβέρνησης θα πρέπει να επικριθεί. Ε, η υπηρεσία για τους πρόσφυγες της, ε, η του για τους πρόσφυγες του ΟΗΕ θα πρέπει να φροντίσει να βοηθήσει αυτούς τους πρόσφυγες εκεί. Θα πρέπει οπωσδήποτε να φροντίσουμε αυτοί οι πρόσφυγες να μπορούν να εγκαταστούν σε τρίτες χώρες. Ευχαριστώ, Μάκλ Κάσμαν. Um, uh ε, ε, καλωσορίζω αυτό το ψήφισμα, αλλά να κάνω την εξή διόρθωση. Δεν πρόκειται για Ισλαμική δημοκρατία, πρόκειται για μια δικτατορία βάρβαρη που χρησιμοποιεί και καταχράται της θρησκείας για τα δικά του συμφέροντα. Αυτή η δικτατορία έχει ως ε, στόχο και μουσουλμάνους και αλλοθρησκούς ε, σιωπούμε βλέποντας ανθρώπους και νέους και παιδιά να απαγχωνίζονται μόνο και μόνο επειδή είναι ομοφιλόφιλοι. και πέραν αυτού το καθεστώς αρνείται πρόσβαση στους ομοφιλόφιλους και σε άλλους ανθρώπους της ίδιας κοινότητα, πρόσβαση στην υγεία, την παιδεία, τις κρατικέ και κοινωνικές πλησίες κλπ. Παρόλα αυτά υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν σε αυτό το καθεστώς και η δική τους ελπίδα θα πρέπει να δώσει ελπίδα και σε εμά. και η δική μας φωνή πρέπει να είναι και η δική τους φωνή. Ευχαριστώ. Κύριο Σταβάρης. Θα περιοριστώ στο να υπενθυμίσω ένα όνομα και να κάνω μια έκκληση. Το όνομα είναι Αμπτουλρέζα Σουμπάς, καθηγητή γιατρό του Πανεπιστημίου των Τυράννων, που επισκέφθηκε το Ιράν και είδε τα θύματα του καθεστώτος. Και στα συμπεράσματά του ανέφερε καθαρά ότι ήταν θύματα βασανισμών. Ο ίδιος δολοφονήθηκε. Το γεγονό ότι γνωρίζουμε πως υπάρχουν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που συνεργάζονται με το Ιρανικό καθεστώς παρεμποδίζοντας ε, τις τηλεοπτικές εκπομπές της αντιπολίτευσης ή δίνοντας software που χρησιμοποιείται στην, στην καταπίεση ε, αποτελεί προσβολή στη μνήμη των νεκρών. Ε, οποιαδήποτε επιχείρηση συνεργάζεται στην ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν θα πρέπει να παίρνει ούτε ένα ευρώ από το κρατικό προπολογισμό και έχουμε βάση δεδομένων μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό να το αποφύγουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει δικαίωμα αυτή τη στιγμή να επιβάλλει χρηματικές ποινές σε εταιρείε οι οποίες με τη δραστηριότητά τους βοηθούν στην παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να ενώσουμε τις προσπάθειές μας έτσι ώστε να αποφύγουμε να παίρνουν χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ. Το ε, καθεστώς αυτή τη στιγμή ε, χτυπάει έτσι γιατί έχει την εντύπωση ότι ε, αδυνατεί ή γιατί έχει την εντύπωση ότι δεν πρόκειται κανένας να ε, του επιβάλλει κυρώσεις. Φαίνεται αυτή είναι η περίπτωση του Ιράν. Κανένας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή στη ΣΥΠΑ δεν ε, προτίθεται να καδεκάσει δημόσια της πράξης αυτού του καθεστώσεως είναι ένα μάθημα για μας. Θα πρέπει να αποφύγουμε διπλά μέτρα και σταθμά ή υποκρισία. Θα πρέπει να ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να τηρούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και στο Ιράν. Δεν μπορούμε να δεχθούμε και να χρηματοδοτούμε εταιρείε που υποστηρίζουν το καθεστώς στη Τεχεράνη. Θα πρέπει να είμαστε πολύ διαφανείς και ξεκάθαροι πάνω σε αυτό το θέμα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα πάντα, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασώσουμε όσους αυτός μπορούμε. Ευχαριστώ κύριο Ρουμπίχ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Εξότιμα ε, επίτροπε. Θα πρέπει να αποφύγουμε να παίρνουμε αποφάσεις έτσι σφαιρικές. Το, ο λαός του Ιράν ε, έχει δικαίωμα να υπάρχει δημοκρατία και θα πρέπει να αναζητήσουμε κατά βάση την ευθύνη ατόμων και να κάνουμε προσφυγή στο ε, ε, δικαστήριο της Χάγης. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα άτομα που είναι υπεύθυνα και αυτά να τιμωρήσουμε γιατί αν επιβάλλουμε κυρώσεις σε όλο το λαό ενδυναμώνουμε τη θέση των ε, εγκληματιών δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό, δεν πρέπει να βάλουμε κυρώσει στους αθώους, αλλά θα πρέπει να έχουμε δικαστική προσφυγή και αποφάσεις ε, κατά εκείνων που καταπατούν το νόμο και θα πρέπει να ενδυναμώσουμε, να υποστηρίξουμε τις δημοκρατικές δυνάμεις στο Ιράν. Θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουν εκείνους που βρίσκονται στο πλευρό μας. Εδώ θα πρέπει να μας δώσετε απάντηση, Επιτροπή. Ευχαριστώ, τελευταίο. κύριο Σκίνερ. Thank you very much, President. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε μεγάλη ευθύνη να σταματήσουμε τις εξαγωγές οποιασδήποτε τεχνολογίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καταπιέσει οποιονδήποτε στον κόσμο, ιδιαίτερα στο Ιράν. Ε, οποιαδήποτε και αν είναι λογισμικό, οποιοδήποτε τύπου. Ε, αν μπορούμε να εντοπίσουμε την πηγή του και αυτό το λογισμικό έχει πηγή στην Ευρώπη, θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σταματήσουμε την εξαγωγή του. Ε, δεν ε, θα δούμε ε, εξεγέρσεις και θανάτους στους δρόμους όπως είδαμε στη Λιβύη. Το Ιρανικό καθεστώς είναι πολύ έξυπνο και δεν θα εκτεθεί με αυτόν τον τρόπο. Είναι πολύ πιο βάρβαρο και ανηλές στη δράση του. Οπότε οποιαδήποτε βοήθεια προς το καθεστώς ακόμα και αν φαίνεται ουδέτερη για την παρακολούθηση διαδηλωτών για παράδειγμα μας καθιστά όλους ενόχους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκύνερη, Επίτροπο κυρία Δαμανάκη. Ακούσατε τη γνώμη των μελών μα, Ποια είναι η άποψη τη Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος της ΥΠΑ της Εκπροσώπου και της Κομισιόν εν γέννη, καλωσορίζω αυτό το ψήφισμα. Θα ήθελα να τονίσω πως ε, η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι φρικτή και επιδεινώνεται. Η καταχρήσεις και οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν χτυπούν όλα ένα και περισσότερο άτομα και οργανισμών και επιδεινώνουν το κλίμα του φόβου και της καχυποψίας. Περασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δικηγόροι, φοιτητέ, δημοσιογράφοι παρανοχλούνται στις φυλακές και πολλές φορές βασανίζονται οι θρησκευτικέ μειονότητες, οι ομοφιλόφιλοι, οι γυναίκες, οι καλλιτέχνες, οι ε, Κινηματογραφιστές επίσης διώκονται. Το Ιράν δεν πληρεί τις διεθνείς του υποχρεώσεις και δεν έχει πουθενά να στραφεί. Οι συχνές συλλήψεις υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δικηγόρων, η διακοπή του ίντερνετ αλλά και η ε, οι υποκλοπές των τηλεφωνικών ε, συνδιαλέξεων οι εκτελέσεις είναι δηληπηρές ε, αποδείξεις αυτών των τάσεων. Θα ήθελα ωστόσο να σας δώσω κάποιες πληροφορίες σε σχέση με τον χριστιανό πάστορα Ιωσέφ Νανταρκάνη, Βρισκόμαστε στην ίδια γραμμή όπως και το Κοινοβούλιο. Το Ιράν πρέπει να ανταποκριθεί στις διεθνές του, διεθνείς του υποχρεώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τον Χριστιανό Πάσταρα. Ζητήσαμε δημόσια την απελευθέρωση του κυρίου Ναδρικάνη και να καταργήσει τις κατηγορίες ε, αποστασίας και παρακολουθούμε την υπόθεση στενά. Επίσης, ε, συμφωνούμε μαζί σας όσον αφορά την δημόσια καταδίκη κράτησης και ε, όπως ο Ζαφάρ Γαναχή και η κυρία Βαφαμέρ. Καλωσορίζουμε την απελευθέρωση της κυρίας Βαφαμέρ, αλλά πολύ ανησυχούμε για το μέλλον της καλλιτεχνικής κοινότητας και της καλλιτεχνικής ελευθερίας. Καλούμε το Ιράν να θέσει μορατόριο στη θανατική ποινή και να σταματήσει όλες τις εκκρεμείς ε, υποθέσεις. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η, η ε, εκτέλεση νεαρών, ανηλίκων. Αγαπητοί κύριοι Ευρωβουλευτέ, ε, δουλεύουμε δραστήρια για να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα για τις ενεργειές μας. Χρησιμοποιούμε την δημόσια ε, διπλωματία. Ο εντυπωσιακό αριθμό δημοσίων δηλώσεων φέτο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα τη κατάσταση. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε το Ιρανικό κοινό, οι δηλώσεις μας μεταφράζονται στα φαρσί και στο ίντερνετ με ενημερώσει από τον το εκπρόσωπο. Στην Τεχεράνη και στι Βρυξέλλε, οι δικέ μα υπηρεσίε συνεχίζουν να παρακολουθούν τι υποθέσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναζητώντα πληροφορίε και διαβιβάζοντα εντόνω τα μηνύματά μα. Η Γενική Συνέλευση του, του ΟΗΕ θα εξετάσει και πάλι φέτο ένα ψήφισμα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν, που ψήφισμα το οποίο ε, υποστηρίζεται ευρύτατα. Θέλουμε επίσης ε, να μπορέσει να πάει στο Ιράν ο δόκτωρ Σαχίμπο, ειδικό ειδικός ε, εισηγητής του ΟΗΕ, του οποίου ο ορισμός έγινε μετά από δική μας πρωτοβουλία. Τον Οκτώβριο φέτος οι Υπουργοί Εξωτερικών μας υιοθέτησαν ένα κατάλογο 61 Ιρανών που είναι υπεύθυνοι για σοβαρές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν είμαστε κατά του Ιρανικού λαού, αλλά Ιρανών, συγκεκριμένων Ιρανών. Ζητήσαμε να παγώσουν τα υπεριοσιακά του στοιχεία και δεν μπορούν να μεταβούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης γνωστοποίησαμε στο Ιράν ότι είμαστε ανοιχτοί για επαφές για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να ολοκληρώσω λέγοντας ότι δυστυχώς δεν υπάρχει καμιά χώρα στον κόσμο που να τραβά τόσο την προσοχή για τα ανθρώπινα δικαιώματα όσο το Ιράν από άποψη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να έχετε καμία αμφιβολία για την αποφασιστικότητά μα να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε να προωθήσουμε και να προστατεύσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Ιράν. Ξέρω πω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμερίζεται αυτή την ανησυχία μα και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ σα ευχαριστώ κυρία Δαμανάκη. Η συζήτηση για την κατάσταση στο Ιράν λοιπόν ολοκληρώθηκε και θα ψηφίσουμε μετά την εξέταση του επο... της επόμενης συζήτησής μας που είναι η Αίγυπτος και συγκεκριμένα η υπόθεση του blogger Αλά Αμπτέλ Φατά. Ο κύριος Καμίνσκι.